Αρχίζουμε λοιπόν, αν συμφωνείτε, σημείο 2 στην ημερησία διάταξη έγκριση αυτής. Σας προτείνω μία τροποποίηση. Γνωρίζετε, το γνωρίζουν όλοι οι συντονιστές και οι σκιώδεις για τις υποχρεώσεις ε, εκφόρτωσης δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε με τον τρόπο που θέλαμε και να το ολοκληρώσουμε εντό τη θητεία αυτή. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα συνεχίσουμε να το συζητάμε και το ε, αφαιρούμε από την ημερήσια διάταξη, διότι δεν προκάνουμε. Εντάξει. Σύμφωνα. Και περνάμε στο επόμενο τρία. Ε, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων, όπω πάντα. Αν έχετε καμιά ερώτηση, διευκρίνηση, θα μα τη διαβιβάσετε για τα πρακτικά. Τέσσερα ανακοινώσει του Προέδρου καμία. Ε, στα διάφορα αν υπάρξει τίποτα. Πέντε, ψηφοφορία. Αλληλευτικές δυνατότητες. Αρχίζουμε αμέσως και πάμε να ψηφίσουμε. Αλληλευτικές δυνατότητες, ε, χρηματική παροχή και ούτω ε, στην Δημοκρατία της Εντάξει, με ανάταση υπέρ Λόβιν. Θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση από τους ε, πράσινους. Ξέρετε ότι αναβλήθηκε η ψηφοφορία για αυτή τη συμφωνία ε, με βάση το άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού γιατί έγινε στρατιωτικό πραξικόπημα και η Επιτροπή, η Επιτροπή θεώρησε ότι θα πρέπει να ισχύσει το άρθρο 96 έτσι ώστε να μην προωθηθούν αναπτυξιακά προγράμματα. Τώρα διενεργήθηκαν εκλογές, αλλά το άρθρο 96 δεν έχει αρθεί ως προς τη Μαδαγασκάρη, γι' αυτό θα απόσχουμε από αυτή την ε, ψηφοφορία. Και ελπίζουμε να αρθεί το άρθρο πριν από την Ολομέλεια. Εντάξει, κυρία Λοβίν, ευχαριστούμε πολύ. Ψηφίζουμε υπέρ. Υπέρ της έκθεσης, κατά, αποχές, 3. Εγκρίνεται. Επόμενο θέμα. Τέσσερις, τέσσερις είναι οι αποχές. Επόμενο θέμα, πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό αλληλευτικών δυνατοτήτων στην Συμφωνία Αλληλευτικές ε, Σύμπραξης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας των Ιθελών. Ε, κάποια παρέμβαση, κάτι, όχι. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, καμία εγκρίνεται. Επόμενο θέμα, το 7, πρωτόκολλο Ευρωπαϊκή Ένωση Κομορών για τι αντιπαροχέ προβλέπων συμφωνία με αλληλευτική σύμπραξη μεταξύ των δύο μερών. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μία τροπολογία η οποία έχει καταπέσει, άρα ψηφίζουμε υπέρ. Παρακαλώ ησυχία. Κατά. Κατά. Αποχές. Λόβιν. Το συγγνώμη κύριε Πρόεδρε που διακόπτω. Αλλά αν θυμάμαι καλά, αποφάσισε η Ολομέλεια ότι στι τελικέ ψηφοφορίε, ακόμα και στι επιτροπέ, θα πρέπει να γίνονται ονομαστικέ ψηφοφορίε. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί απλώ το κάνουμε για να τι χειρό. No, eh, το λέω Θέλουμε να δούμε τις ψήφους, ε, γιατί ε, δυστυχώς ε, δεν λειτουργεί, δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Γι' αυτό το λόγο. Μόνο γι' αυτό το λόγο, όχι επειδή θέλω εγώ να κάνω το αντίθετο. Εγώ πάντα ακολουθώ τον κανονισμό. Αν θέλετε τώρα μπορούμε να το κάνουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε αυτό το σημείο το 7. Αρχίζει η ψηφοφορία. Esa αυτό ήταν ο λόγο. Πέρασε. Α, δεν λειτουργεί. working. Μερικών ε, λειτουργεί, άλλων όχι. Cámbiate, María, ε, comienza de Λοιπόν, αρχίζουμε και πάλι. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία τώρα. Πέρας. 15 ψήφοι υπέρ. Κανείς δεν αντιτάσσεται καμία αποχή. Εγκρίνεται. Λοιπόν, επόμενο σημείο 8. Έκθεση Τόμας για τη Διεθνή Σύμβαση του Διεθνούς ε, Ναυτιλιακού Οργανισμού. Ε, ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με ομοφωνία. Ψηφίζουμε την εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε σχέση με την έκθεση Ρωμέβα. για την αδήλωτη παράνομη και λοιπά. Λοιπόν, πέρας, ε, ομοφωνία, τέλος, ε, επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το 9, ε, τον προπολισμό 2015, εισηγητής ο κύριος Γκάλαχερ, έχετε το λόγο. Σημείο 10. Πατ. Πατ. Πατ. We are waiting for you. Is your point? it. Go ahead. Stuart. Chairman, the members, if they haven't, should have. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε διανέμει, έχουμε, έχουμε διανέμει στα μέλη μια επιστολή που είναι αυτή που αναφέρεται το ζήτημα. Θα ήθελα να ζητήσω από τα μέλη να την διαβάσουν. Αν τυχόν δεν την έχουν θα τους ε, έρθει σύντομα, θα τη λάβουν σύντομα και εάν θα ήθελαν να την τροποποιήσω κατά κάποιον τρόπο και επιμένουν σε αυτό, να μου το πούν ευχαρίστως θα το κάνω. Πάντω, θα έλεγα κύριε Πρόεδρε ότι είναι πολύ τυποποιημένη επιστολή και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ε, το συζητήσουμε και πολύ. Πάντως εάν κάποιο μέλο θα ήθελε να την τροποποιήσει αυτήν την επιστολή Ευχαριστώ. Okay, thank you very much indeed. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γκάλαχερ, πράγματι τα μέλη άκουσαν αυτό που ζητήσατε. Εάν έχουν οποιοδήποτε σχόλιο, να το στείλουν. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μας ε, χρειάστηκε να πάει στην Επιτροπή Γεωργίας για να ψηφίσει. Γι' αυτό ανέλαβα την Προεδρία. Η Επιτροπή μου πως θέλει το λόγο να σχολιάσει. Όχι. Κάποιο μέλος, κάποιος βουλευτής. Όχι. Επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης εκτός αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Κύριε Γκάλαχερ, ναι. Ναι, ήθελα να πω ότι μιας και είναι εδώ η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήταν σκόπιμο να ακούσουμε την άποψή της. Ο Πρόεδρος, ναι, αλλά νομίζω δεν είναι εδώ. Κανένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί προχωρήσαμε γρήγορα στην ημερήσια μας διάταξη. Ωραία. προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω τις σημειώσεις του Πρόεδρου που ήταν στα Ισπανικά και φαίνεται ότι μάλλον πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα που είναι παρουσίαση από το θεματικό τμήμα Β για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στην Αλία. Έχουν έρθει εκπρόσωποι της, ε, που θα μας παρουσίασαν αυτό, αυτό το θέμα. Όχι, έχουμε προχωρήσει πολύ γρήγορα. Υπάρχει μια... Υπήρξε μάλλον το πρωί μια ε, παρατηρημένη συζήτηση για το ζήτημα της ε, απαγόρευσης εκφορτώσεων. Φαίνεται λοιπόν ότι πρέπει να περιμένουμε και πρέπει να διακόψουμε τη συνεδρίαση μέχρι να έρθουν οι εκπρόσωποι της Corporate Solutions που θα μας κάνουν αυτή την παρουσίαση. Ζητώ συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Καλαχέρ, να προτείνω, μιας και θα έρθει η Επίτροπος στις 12. Αν ξεκινήσουμε τη συζήτηση 11.30, νομίζω θα έχουμε χρόνο αρκετό στη διάθεσή μας, ο Πρόεδρος. Άρα μου ζητάτε να ζητήσω την Επίτροπο να έρθει στις 11.30, αυτό μου ζητάτε. We deal with the item perspectives for the development of tourism activities. Όχι, όχι, άλλο λέω. Οι προοπτικέ για την ανάπτυξη τουριστικών διαστηριοτήτων στην Αλγία, αυτό να το συζητήσουμε στι 11.30. Για να μην χρειαστεί να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα και ένα διάλειμμα μετά. Ο πρόεδρο. Η πρόταση λοιπόν του κυρίου Γκάλαχερ είναι να συζητήσουμε την παρουσίαση στι 11.30. Δηλαδή να συζητήσουμε το θέμα 11 στις 11.30 για να μην χρειαστεί διάλειμμα ανάμεσα στο θέμα 11 και στη συζήτηση με την Επίτροπο. Συμφωνούμε. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έρθουμε εδώ στις 12 για να συζητήσουμε με την Επίτροπο. Okay, is that agreed then that we adjourn until 11? Ωραία, συμφωνήσαμε λοιπόν. Διακόπτουμε έως τις 11.30 έρθουμε στι 11.30 και επί μισή ώρα θα συζητήσουμε τις προοπτικέ για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Ελία και στις 12 θα έρθει η ε, Επιτροπό, Η κυρία Λεβίν. Ε, είμαστε σίγουροι ότι μας φτάνει μισή ώρα για την παρουσίαση και τις ερωτήσεις. Μπορείτε να ήταν καλύτερο να δώσουμε 45 λεπτά. 11 και 4. Εντάξει. Άντε, 11 και 4. Διακόπτουμε τη συνεδρίαση μέχρι τι 11 και 4. Γεια σα.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 Λοιπόν, συνεχίζουμε παρακαλώ μετά από το διάλειμμα. Νομίζω ότι φαίνεται ότι βαίνουμε προς το τέλος της θητείας. Καλά είναι να προεδρεύει ο συνάδελφος Στρούαν Στίβενσον γιατί τα διεκπεραιώνει πολύ πιο γρήγορα από μένα. Και μας έμεινε μεγάλο διάλειμμα για καφέ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Στίβενσον. Πριν περάσουμε όμως στο σημείο 11, μου έλεγαν ότι ξεχάσαμε να πούμε ότι η πρόταση κανονισμού για τα ε, τυχαίες ε, αλλιεύσεις κοιτοδών ε, έχει αλλάξει προθεσμία. 19 Απριλίου στις 12 Μαρτίου, συγγνώμη, αύριο δηλαδή, 19 Μαρτίου στις 12. σημείο 11 λοιπόν, η παρουσίαση για τις προοπτικές ανάπτυξης των τουριστικών ε, δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αλληλεία. Είναι από το θεματικό τμήμα Β. Το ενημερωτικό σημείωμα ανατέθηκε στην Corporate Solutions. Δεν θα σας πω εγώ περί τίνος πρόκειται. Θα δώσουμε αμέσω το λόγο καλύτερα ε, για να μην χάσουμε χρόνο στον κύριο Γιούλιους Φούστερ της Corporate Solutions και θα έχουμε γύρω στα 20 λεπτά για να μας παρουσιάσει το ενημερωτικό σημείωμα και στη συνέχεια να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές που θα το επιθυμήσουν. Παρακαλώ κύριε Φούστερ. Και καλωσορίσατε βεβαίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας. Ε, θα σας κάνω την ε, παρουσίαση στα ε, αγγλικά. Είναι και διαφάνεια στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Το ζήτημα είναι εξαιρετικά ευρύ. Θα ξεκινήσω από το γενικότερο και θα εξειδικεύσουμε αργότερα κατά τη διάρκεια των 20 λεπτών της παρουσίασης. Το ζήτημα της αξιοποίησης της αλίας για τον τουρισμό και τις διάφορες διάφορους τομείς στους οποίους τέμνονται οι δραστηριότητες της αλίας και ο ε, τουρισμός, ο τουρισμός με σκοπό την αλία. Μετά Έχουμε 7 μελέτες περίπτωσης και βέλτιστες πρακτικές που θα ήθελα να σας παρουσιάσω. Όπως γνωρίζετε πολλά προγράμματα ήδη έχουν ξεκινήσει. Υπάρχουν πάνω από 6.000 γαλάζιες σημαίες και προσπάθησα να καλύψω προγράμματα από διάφορες περιοχές της Ευρώπης, στο βορρά, στο νότο, ανατολικά και δυτικά. Και τέλος θα κλείσω με κάποιες, κάποια διδάγματα που αποκομίσαμε. Έχουν διεξαχθεί διάφορες μελέτες για τη σχέση τουρισμού και αλίας τα τελευταία 15 χρόνια. Ξεκίνησε με ένα εργαλείο προσανατολισμού και το πρώτο ταμείο για την αλία ακολούθησε και στην επόμενη προγραμματική περίοδο έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας. Όπως σας είπα, έχουμε επιλέξει σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Β ορισμένες μελέτες περίπτωσης, προσπαθώντας να καλύψουμε όλων των ειδών τα έργα, μικρά ή μεγάλα ε, προγράμματα ή ε, σκάφη στο βορρά, στο νότο, σε διάφορες περιοχές. Εγώ θα σας παρουσιάσω ορισμένα από αυτά. Δεν χρειάζεται εγώ να σας εξηγήσω ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της Αλίας σήμερα. Εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα. Αυξάνεται το κόστος, αυξάνεται το κόστος το εργατικό, ε, για τα εργατικά για τους ε, αλληλείς, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται και τα αλληλευτικά αποθέματα. Γνωρίζουμε ότι η αλληλευτική δραστηριότητα συγκεντρώνεται σε ορισμένε χώρε, κυρίω στην Ισπανία, τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τι κάτω χώρε, τη Ολλανδία, αλλά βέβαια και άλλε χώρε όπω η Πολωνία και νέα κρατημέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και εκείνα τα νέα κρατημέλη αντιμετωπίζουν πολλέ δυσκολίε προσπαθώντα να βοηθήσουν τις κοινότητες αλλιέων τους να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον. Όπως είπα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηρίξει τον κλάδο της Αλίας από το 2000, αρχικά με τις προσπάθειες ε, διαφοροποίησης. Υπήρχε ο άξονας 4 στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αλία από το 2007 στο 2013, στο πλαίσιο του οποίου ε, κατανεμήθηκαν 4 δισεκατομμύρια 304 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία σχεδόν στο σύνολό τους χρησιμοποιήθηκαν για τη διαφοροποίηση, για την βελτίωση ε, της ηχθειοκαλλιέργειας και άλλων τομέων. Και στο πλαίσιο της διαφοροποίησης, ένας σημαντικός τομέας ήταν ο τουρισμός, η σύνδεση της Αλίας με τον τουρισμό. Και θα δείτε και αργότερα στην παρουσίαση, είναι αυτός ο οποίος ε, συγκέντρωσε και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις τοπικές κοινωνίες της παράκτειας. Φυσικά αυτό εντάσσεται σε μια γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές, του θαλάσσιου τουρισμού. Και όπως γνωρίζουμε, 6,5 δισεκατομμύρια στην, έχουν προβλεφθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο, δηλαδή μέχρι το 2020, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Όπως βλέπετε στο διάγραμμα, οι περισσότερες θέσεις εργασίας βρίσκονται στον Ατλαντικό κενό και, στον, ε, και στη Μεσόγειο. Φυσικά στη Μεσόγειο η απασχόληση στον τουρισμό είναι πολύ πιο μεγάλη, ενώ στον Ατλαντικό προφανώς οι θέσεις εργασίας αφορούν περισσότερο την αλία παρά τον τουρισμό. Βέβαια τα πράγματα εξελίσσονται. Αυτό που σας δείχνω εγώ τώρα είναι μια ε, φωτογραφία, μια απεικόνηση της κατάστασης όπως είχε τότε. Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορούμε να ορίσουμε τον τουρισμό. Πρώτα απ' όλα τον τουρισμό που συμπεριλαμβάνει και μετακίνηση, που καλύπτει 7 έως 15% ανάλογα με το, εάν, με το ποιος τον μέθρα. Αλλά αν συνυπολογίσουμε και όλες τις παρελκόμενες υπηρεσίες, τους, υπηρεσίες τους ε, διάφορους ε, άλλους κλάδους που δραστηριοποιούνται που υποβοηθούν τον τουρισμό, ε, είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των απασχολούμενων στον τομέα συνολικά και γι' αυτό ενδιαφέρει τις τοπικές κοινωνίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποστηρίξει μέσω του άξονα 4 πολλά ε, προγράμματα. Πρώτα απ' όλα δημιουργήθηκαν τα flags, οι τοπικές ομάδες δράσης ε, για την αλία και αργότερα αυτές εντάχθηκαν στο δίκτυο Farnet ξεκίνησαν δειλά-δειλά, αλλά τώρα σιγά-σιγά αναπτύχθηκε και ορίμασε, θα έλεγα, το πρόγραμμα αυτό. Μάθαμε από τα λάθη μας στο παρελθόν, τους έγιναν και κάποιες αξιολογήσεις αντικτύπου. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ειδικό στον τομέα του τουρισμού και της αλίας, ασχολούμαι γενικά με την οικονομική ε, ανάπτυξη. Θα έλεγα λοιπόν ότι χρειάζεται να γίνουν ακόμα περισσότερες αναλύσεις και ακόμα περισσότερες μελέτες αντικτύπου για να δούμε πώς μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να αυξηθεί το εισόδημα των αλλιών και πώς θα βοηθήσουμε τις τοπικές κοινότητες ε, αλλιέων. Όπως σας έλεγα λοιπόν, 6 ε, δισεκατομμύρια, 400 εκατομμύρια ευρώ έχουν προβλεφθεί για την επόμενη προγραμματική περίοδο στο πλαίσιο του δικτύου Farnet. Στο παρελθόν τα χρήματα αυτά αφορούσαν, είχαν μάλλον αποδοθεί κυρίως σε χώρες όπως η Ισπανία, η Πολωνία, οι κόκκινες γραμμές που βλέπετε στο διάγραμμα στην οθόνη σας. Οι μπλε γραμμές αντιπροσωπεύουν το συνολικό ποσό του ε, Ταμείου για την Αλία. Βλέπετε λοιπόν ότι στην Πολωνία ε, ε, αποδόθηκαν περισσότερα χρήματα γιατί είχε περισσότερες προκλήσεις να αντιμετωπίσει. Είχε μεγαλύτερη δουλειά να κάνει στον τομέα, για παράδειγμα, ε, της, ε, του επαναπροσανατολισμού των τοπικών αλληλευτικών κοινοτήτων. Αυτά για το παρελθόν. έχουμε αυτή την τυπική εικόνα ενός γραφικού λιμανιού και αν έχει ομορφές βαρκούλες ακόμα καλύτερα. Αλλά ο τουρισμός και η σύνδεση του τουρισμού με την αλληλεία έχει πάει πολύ πιο μακριά. Υπάρχει προφανώς ο τουρισμός στις παράκτης περιοχές που χρειάζεται να αναπτυχθούν και οι υποδομές στην ενδοχώρα για τη φιλοξενία, για στο λιμάνι, για να υποστηριχθεί η άφηξη των τουριστών, αλλά υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα ο, η, διάφορα φεστιβάλ αλλά ταυτόχρονα αναπτύσσεται σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Φινλανδία και ένας τουρισμός αλληλευτικός στην ενδοχώρα. Ο τομέα που έχει μελετηθεί περισσότερο και για τον οποίο γνωρίζουμε τα περισσότερα εξαιτία των αδιωτηρωτήτων του είναι ο λεγότερος ε, τουρισμός αλίας, pesca tourism στα αγγλικά. Όταν το χρησιμοποιούσαμε όμω αυτό τον όρο κανείς δεν τον καταλάβαινε παρά το γεγονό ότι είναι ο επίσημος όρο που χρησιμοποιεί το Farnet. Εάν κανεί μιλήσει με του ταράδε, και τους πει πες μου του λένε τι ε, είναι ένας ε, όρος που χρησιμοποιεί η Επιτροπή και αναφέρεται στον τουρισμό δηλαδή όταν ο επισκέπτης ανεβαίνει πάνω στη Ψαρόβαρκα μαζί με τους αλληλείς και μαθαίνει πώς γίνεται η αλληλεία και τους παρακολουθεί καθώς εργάζονται. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ως δραστηριότητα γιατί δίνεται τη δραστηριότητα στου τοπικού αλληλεί απλώ να συνεχίσουν τη δουλειά του ω συνήθω και ταυτόχρονα να υποδεχθούν και τουρίστε, χωρί να σταματήσουν να ψαρεύουν. Επίση, βοηθάει έτσι ώστε το κοινό ε, μέσω του τουρισμού να ευαισθητοποιηθεί και να γνωρίσει καλύτερα και στον κόσμο της αλίας που είναι πολύ ιδιαίτερος. Πολύ συχνά ε, παραγγέλνουμε ένα ψάρι και δεν γνωρίζουμε από πού έχει έρθει, δεν γνωρίζουμε πώς πώς γίνεται το, το ψάρεμα, δεν γνωρίζουμε τίποτα από όλα αυτά. Και ο τουρισμός αλίας δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει και τις δυσκολίες, το πόσο ε, δύσκολες είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι ψαράδες ε, με την υγρασία στη θάλασσα, το δουλεύουν 16 ώρες, είναι ένας τομέας στον οποίο είναι αδύνατο για παράδειγμα ε, ένας ανήλικος να, να εργαστεί. Εξηγείται επίσης και το, το γεγονό ότι η μείωση των αλλιευτικών αποθεμάτων δημιουργεί προβλήματα στους αλληλείς, αλλά με τον τουρισμό μπορούν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Όπως γνωρίζετε, εάν το εισόδημα κάποιου βασίζεται μόνο από την αλληλεία είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, μειώνεται τα αποθέματα, ενώ με τον τουρισμό, τουρισμό μπορεί να το αντιμετωπίσει. Ωστόσο, σε ένα πιο θεσμικό επίπεδο, στο επίπεδο της οργάνωσης αυτής της διαδικασίας από το κράτος, υπάρχει κενό. Δεν είναι διαφανές, αλλά ε, στο ενημερωτικό σημείο υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο στις διάφορες χώρες. Βασικά μόνο μία χώρα έχει μια νομοθεσία από το 1999 για τον ε, τουρισμό αλίας, η Ιταλία, ε, η οποία νομοθεσία ορίζει με βάση ποιους όρους μπορεί μια, ε, ε, ένα σκάφος να δεχθεί τουρίστες. Στη Γαλλία υπάρχει μία απαλλαγή από το ΦΠΑ ειδικά για τις τους, αλείς που υποδέχονται τουριστές. Ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο αξιολογούν, έχει εγκριθεί η νομοθεσία και αναμένονται τα εκτελεστικά μέτρα μετά το πιλωτικό πρόγραμμα. Στην Ισπανία, στην Καταλωνία και στην ε, Γαλλικία έχουν περιφερειακή νομοθεσία. Σε άλλες περιοχές όπως τη Βαλένθια υπάρχει ενδιαφέρον για να γίνει κάτι παρόμοιο. Εξετάζεται επίση και το ενδεχόμενο στην Ισπανία να εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο νομοθεσία, αλλά δεν έχει γίνει κάτι το ακόμα. Στην Κύπρο έχει ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα, στην Φιλανδία επίση, σε άλλε 8 χώρε. Δεν απαγορεύεται, αλλά ταυτόχρονα επιβάλλονται ε, τα μέτρα που ισχύουν σχετικά με τις μεταφορές γενικά. Που είναι πολύ αυστηρά το οποίο στην, στην πράξη σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο δεν μπορεί στην πράξη ε, να γίνει. Στις χώρες εκείνες δηλαδή που δεν έχουν συγκεκριμένη νομοθεσία δεν γίνεται. Στη Βουλγαρία, στη Γερμανία, στην ε, κάτω χώρες, στην Ιρλανδία, στην Σλοβενία, σε 8 χώρες απαγορεύεται. Ρητά. Απαγορεύεται σε ένα σκάφος που ψαρεύει να ε, έχει και επιβάτες τουρίστες. Μπορεί να υπάρχει ένα άλλο σκάφος που να ακολουθεί το αλλιευτικό και να παρακολουθούν από εκεί οι τουρίστες, αλλά αυτό δεν είναι ικανοποιητικό. Επομένω, όπως βλέπετε, η νομοθεσία διαφέρει πολύ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και χρειάζεται εναρμόνιση. Υπάρχει επίσης πληθώρα περιφερειακών, τοπικών κανόνων και τοπικής νομοθεσίας. Στην πραγματικότητα μόνο ε, η Ιταλία, η Γαλλία και αυτές οι τοπικές κοινότητες που σας ανέφερα έχουν νομοθεσία και είναι εύκολο να γίνει μια διαπραγμάτευση μεταξύ αυτών των πέντε. Αλλά υπάρχει ίσως αυτή η αίσθηση ότι το ζήτημα αυτό αφορά μόνο τις χώρες του Νότου αλλά όπως καλά γνωρίζετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ισχύει αυτό. Όλα τα κράτη-μέλη θα, θα, θα συμμετείχαν σε μια τέτοια διαπραγμάτευση και μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι οι Έλληνες, γενικά οι Ιταλοί, οι νότιες χώρες θα είχαν μια άλλη προσέγγιση ενώ οι Δανείοι και οι βόρειες χώρες μια άλλη. Σε όλες, ορισμένες περιοχές διαφέρει η ονομασία που δίνεται στον αλληλευτικό τουρισμό και κάποιοι συμπεριλαμβάνουν και δραστηριότητες τουριστικές στην ξηρά. Μια έτσι, εστιατόριο που πουλάει ψάρι ή όλες αυτές, όλα αυτά τα παρεμφερεί. Θα έλεγα λοιπόν ότι το τομέα είναι κάπως ετερογενής. Δεν υπάρχει ένα και μοναδικό επιχειρηματικό μοντέλο ή ένας τρόπος για να αναπτυχθεί μια αλληλευτική κοινότητα. Φυσικά θα μου πείτε, κάθε τοπική κοινότητα είναι διαφορετική, διαφέρουν τα ψάρια και το αλληλευτικό απόθαμα, μα διαφέρει η λογική, η φιλοσοφία, οι τοπικές εδρατεραιότητες, επομένως δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένα ενιαίο και μοναδικό μοντέλο. Δεν λέω αυτό. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να υπάρχει ένα πλαίσιο ένα πλαίσιο για ένα επιχειρηματικό μοντέλο, στο πλαίσιο του οποίου ο καθένας μετά θα μπορούσε να εξειδικεύει με βάση τις τοπικές συνθήκες. Γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα υποδομής, όπως για παράδειγμα η πρόσδεση των πλοίων, τα GPS που χρειάζονται υποδομές στο λιμάνι και κάποια άλλες, κάποιες άλλες δραστηριότητες που θα τις ονόμαζα soft, που είναι η προώθηση, που είναι ο τρόπος με τον οποίο διαφημίζεται ο τουριστικός προορισμός. Ας περάσουμε τώρα σε άλλους συναφείς τομείς, όπως τον θαλάσσιο τουρισμό ή την άλλη αναψυχής. Εδώ χρησιμοποίησαμε διεθνώς παραδεκτούς ορισμούς. Η αλία αναψυχή όπως γνωρίζετε έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές φορές και έχουν υπάρξει και ας πούμε κάποιες εντάσεις, κάποια προβλήματα μεταξύ τους επαγγελματίες παραδοσιακούς ψαράδες και εκείνους που ψαρεύουν μόνο για λόγους αναψυχής. Η Επιτροπή Αλίας δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα γιατί είναι δύσκολο να, βρει μια, να βρεθεί ένα συμβιβασμό ανάμεσα στου ερασιτέχνε ψαράδε και του επαγγελματίε. Ο ΦΑΟ και άλλοι διεθνεί οργανισμοί το έχουν μελετήσει αυτό το θέμα και έχουν πει ότι για παράδειγμα θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των παράπλευρων ελευμάτων από τους ερασιτέχνες ή τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργούνται στο οικοσύστημα από την αερασιτεχνική αλία. Αυξάνεται ο τομέας, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δαπανίσει και πολλά κονδυλία για να ενισχύσει την αερασιτεχνική αλία. Θα έλεγα ότι ήταν μάλλον κάποια μικρά προγράμματα στην Βουλγαρία, στη Σουηδία και αλλού και άλλοι ανέλαβαν πρωτοβουλίες όπως η Φινλανδία, αλλά περισσότερο για να αναλύσουν τι αντίκτυπο έχει η, η, η, η αλία αυτή, όχι τόσο η ερασιτεχνική όσο περισσότερο η αλία στην ενδοχώρα. Θαλάσσιος τουρισμός. Και πάλι εδώ οργα, ε, ακολουθούμε τον ορισμό του ICTMS, ο οποίος συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε μετακίνηση, στην οποία τελικά καταλήγουμε σε μια περιοχή θαλάσσια ή παράκτια. Επομένως εδώ είναι, μιλάμε για κάτι πολύ γενικότερο, θα συμπεριλαμβανόταν η αλληλεία, ο, ο, ο τουρισμός, αλλά επίσης και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα στην ξηρά, για παράδειγμα ένα φεστιβάλ, ένα, μια εκδήλωση ή μια επίσκεψη με ξενάγηση σε μια ψαραγωγορά ή ένα μουσείο για τα απειλούμενα είδη ή ένα μουσείο φυσικής ιστορίας, όλα αυτά. Όλες αυτές τις δραστηριότητες τις εντάσσουν στο πλαίσιο της χαλάζιας οικονομίας που έχει απασχολήσει και την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει θεωρηθεί θέμα προτεραιότητας πρόσφατα και σίγουρα αναμένουμε ότι στο επόμενο, στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα υπάρχουν αρκετά χρήματα στον τομέα αυτό, στον, στον άξονα 4. Ελπίζουμε όλοι ότι αυτή η γαλάζια ανάπτυξη θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και μιλάμε εδώ για φεστιβάλ, για ε, αξιοποίηση ιστορικών ε, χώρων που θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να προωθήσουν την αλία. Μιλάμε επίσης για ξεναγήσει σε θαλάσσιους ε, ε, προορισμού. Πρόσφατα στο Τρινιδάδι είχα πάει σε μια ξενάγηση κοραλιογενείς υφάλους. Όλα αυτά τέλο πάντων εντάσσονται στον τουρισμό το θαλάσσιο. Φυσικά όλα εξαρτώνται από το, το, το φυσικό περιβάλλον κάθε περιοχής. Χρειάζεται να έχει κάτι ελκυστικό για να προσελκύσει τουρίστες. Όμως το σημαντικότερο είναι, για, κατά την άποψή μου, η καινοτομία. Πρέπει να υπάρχει κάτι ξεχωριστό για να πάνε εκεί οι τουρίστες. Γι' αυτό πιστεύω ότι τα flags και οι διάφορες κοινότητες που συμμετέχουν σε αυτά έχουν μεγάλη σημασία. Αλλά φυσικά πρέπει κανείς να είναι και προσγειωμένος. Δεν είναι δυνατόν να περιμένει ότι ένα εκατομμύριο επισκέπτες θα έρθουν μόνο και μόνο επειδή άνοιξε ένα μουσείο για το ψάρεμα. Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργηθούν άνθρωποι με ειδίκευση, με γνώση στον τομέα του τουρισμού, της φιλοξενίας. Αυτό δεν είναι απλό, δηλαδή δεν είναι εύκολο κάποιο ο οποίο είναι επαγγελματίας, αλλιέας, ε, ξαφνικά να γίνει ξενοδόχος ή να μάθει πώ να αντιμετωπίζει τον τουρισμό. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς ε, θα βοηθήσουμε και θα δώσουμε δυνατότητες εκπαίδευση και ε, κατάρτισης στη νέα γενιά. Ας κοιτάξουμε, κοιτάξουμε τώρα τις μελέτες περιπτώσεων, τις βέλτιστες πρακτικές που ήθελα να σας παρουσιάσω. Ε, έζησα κάποια χρόνια στην ε, Καταλωνία και πρέπει να σας πω ότι είναι... Ε, ζητώ συγγνώμη από τους Ιταλούς ε, πρωτοπόροι στον τομέα του ε, τουρισμού του ελευτικού στη Βαρκελόνη και σε άλλες περιοχές της Καταλωνίας είχαν διάφορες επιτυχίες οι μόνοι που προσπάθησαν όμως να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο ήταν η Ιταλία. Και το συμπέρασμα ήταν ότι στην Ιταλία η... Συμπέρασμα ήταν ότι αν αυξηθεί ο ε, ο, αν, αν αυξηθεί ο αλληλευτικό τουρισμό, οι ψαράδε θα μπορέσουν να μειώσουν τι ώρε εργασία του από 16 σε 11 και την ε, το ημερήσιο ελίευμα κατά 2 έω 5 κιλά. Βέβαια αυτό ήταν μια συγκεκριμένη μελέτη αντικτύπου που θα χρειαζόταν να κάνουμε και άλλες, σε άλλες περιοχές. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο ακόμα, ούτε ήταν δύσκολο μάλιστα να βρούμε και αυτήν την μία μοναδική μελέτη αντικτύπου στο Φάρνετ. Θα επιταχύνω λίγο γιατί δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Στη Φιλανδία προσπάθησαν να αποσωτικοποιήσουν, να μετρήσουν τον αντίκτυπο που έχει ο αλληλευτικός τουρισμός στην ενδοχώρα. Αλλά αυτό που μας λένε είναι δύσκολο να το μετρήσουμε αυτό γιατί δεν έχουμε έναν ξεκάθαρο ορισμό ε, του αλληλευτικού τουρισμού. Θα χρειαστεί να, να, να καταμετρώνται για παράδειγμα ε, όταν ένα λιευτικό σκάφος υποδέχεται τουρίστες και κάνει, μια, και κάνει ένα τουρ. Πάω στην Ιταλία για το φεστιβάλ ε, Αλίας Τόνου. Και εδώ διαπιστώνουμε τη σημασία της υποδομής. Αν δεν υπάρχουν υποδομές, αν δεν υπάρχουν οδικοί άξονες που να οδηγούν εκεί που γίνεται το, αυτή η εκδήλωση, υπάρχει πρόβλημα. Συνήθως λοιπόν σε μια τουριστική περιοχή πρέπει πρώτα να φροντίσει κανείς. Να, να, να ξεκινήσει με κάτι μικρό και σιγά σιγά να το ενισχύσει. Όπως σας είπα λοιπόν η κατάρτιση είναι πολύ σημαντική. Αν μιλούμε για ψαράδες πρέπει να απευθυνθούμε στους γιους τους, στους ανεψιούς τους, στις συζύγους τους για να μάθουν πώς να ασχολούνται με όλα αυτά. Και επίσης χρειαζόμαστε και ένα, ένα σχέδιο. Δεν αρκεί απλώς ένα σεμινάριο. Χρειάζεται όλη αυτή η κατάρτιση να εντάσσεται σε ένα πλαίσιο. Που τελικά να επιτρέπει στους ψαράδες να διαφοροποιήσουν τις υπηρεσίες που τελικά παρέχουν. Και χρειαζόμαστε, όπως για οποιοδήποτε προϊόν, να υπάρχει κάτι που να το ξεχωρίζει, να το διαφοροποιηθεί από όλα τα άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα. Και για την προώθηση χρειάζεται η αξιοποίηση και των παραδοσιακών αλλά και των νέων μέσων. Τα νέα μέσα, ίντερνετ λοιπά, σήμερα καλύπτουν το 90% των, ε, του, του marketing για τον τουρισμό. Όταν όμως μιλάμε για μια μικρή κοινότητα αν έχουμε ένα μικρό ξενοδοχείο στην Κατάρα, στην Ιταλία, δεν θα... Τσετάρα, συγγνώμη, στην Ιταλία, ε, οι υπηρεσίες δεν είναι σε θέση να υποδεχθούν εκατοντάδες τουρίστες και πολύ συχνά τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα και ε, μέσω μιας ηλεκτρονικής καμπάνιας προώθησης μπορεί κανείς να βρεθεί σε μια θέση να μην μπορεί να αντιμετωπίσει όλους αυτούς που τουρίστες θα, θα έρθουν και αυτό ε, μπορεί στην πραγματικότητα να οδηγήσει σε αντίθετο αποτέλεσμα, να, να, να, υπονομεύσει την προσπάθειά του, να έρθουν τόσο πολλοί που να μην τα καταφέρει και να δημιουργήσει κακό όνομα. Από μόνη της μια τοπική κοινότητα δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά. Να, τελειώνεται σιγά σιγά, ολοκληρώνεται, να γίνει και καμιά συζήτηση. Επίσης, ε, η μεγάλη σημασία έχει ο ρόλος των γυναικών και των ε, γιών τους. Ε, δηλαδή, οι γυναίκες επιχειρηματίες όχι μόνο να βοηθήσουν στο εστιατόριο και να μαγειρεύουν να ανοίγουν την επιχείρηση. Μπορούν να κρατάνε τα λογιστικά βιβλία γιατί ο άντρας δεν θα το κάνει, ο σύζυγος δεν θα το κάνει. Επίσης η εποχικότητα, τα φεστιβάλ, τα μουσεία, το ότι πρέπει να κάνουμε κάτι εκτός σεζόν είναι πολύ σημαντικό. Η επιστημονική κοινότητα θα πρέπει να βοηθήσει έτσι ώστε οι ε, αλληλείς να δίνουν τις πρώτες πληροφορίες για τα αλλιεύματα, τα προβλήματα στις οικολογικές περιοχές, ε, αν διαπιστώσουν ε, μολύνσεις κλπ. Επίσης το περιβαλλοντικό, η καθαρή προορισμοί, για να τους κατονομάσουμε έτσι, και αυτές οι νέες τουριστικές δραστηριότητες στρέφονται ε, προς ε, τους ε, νέους που στρέφονται προς την οικολογία έτσι ώστε οι οικογένειες με τα παιδιά να πηγαίνουν σε προορισμούς, σε καθαρούς προορισμούς, χωρίς μολύνσεις και ούτω καθεξής. Με συγχωρείτε που χρειάστηκε να μακρηγορήσω, τα άλλα θα τα βρείτε στις σημειώσεις μου. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, σπουδή με την οποία έπρεπε να μας παρουσιάσετε την εισήγησή σας. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στους βουλευτές, ποιοι θα ήθελαν το λόγο για να σχολιάσουν. Τόμας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και σας ευχαριστούμε πολύ για την ε, εισήγησή σας. Έχω μία σειρά σχολείων και ερωτήσεων. Μιλάτε για την γαλάζια ανάπτυξη και την γαλάζια οικονομία. Μιλήσατε για 7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ε, ε, είναι τα στοιχεία που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν πρόκειται για δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ε, τουρισμό, σχετίζονται με τις ανανεώσιμες και τη θαλάσσια βιοτεχνολογία. Έχετε κατά προσέγγιση στοιχεία έτσι ώστε να δούμε σε αυτή τη γαλάζια ανάπτυξη πώς έχουν οι εξελίξεις και ποιες είναι οι προοπτικές, ποιες θέσεις εργασίας αφορούν τον τουρισμό στην γαλάζια ανάπτυξη. Δεύτερον, όπως είπατε, ο τουρισμός είναι πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα για τα παράκτια μας, αλλά έχει εποχικό χαρακτήρα. Η αλία όμως και οι άλλοι ε, τομείς που αφορούν τεχνολογικά ζητήματα και άπτονται της αλληλείας επιτρέπουν βιώσιμες θέσεις εργασίας και σταθερές, όχι εποχικές. Τέλος, τελευταίο σχόλιο ή ερώτηση. Μιλήσατε για την αναγκαία εναρμόνιση μεταξύ της αλίας ε, αναψυχής της εραστεχνικής αλίας ε, με την επαγγελματική. Θα πρέπει να συνδέσουμε την κοινή πολιτική αλίας με ένα βιώσιμο σχήμα. Όμως, όσο αφορά την τουριστική αλία, δεν υπάρχει αυτή η υποχρέωση ε, ποσοστώσεων, ας πούμε. Εκτός από ορισμένε εξαιρέσεις, αυτό θα γενικευθεί για ολόκληρη την αλία. Θα, δώσουν το λόγο, θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους ε, βουλευτές και μετά θα μπορέσετε να απαντήσετε. Λαβίν. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για την παρουσίαση και τη μελέτη. Είναι πρόσδεκτα τα θετικά στοιχεία για τα προγράμματα του άξονα 4 Πιστεύω ότι το δημόσιο χρήμα θα πρέπει να δαπανάται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το δημόσιο καλό. Και νομίζω ότι τα αριθμητικά σας στοιχεία και η ανάλυση σας δείχνουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον τουρισμό και για τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Έχουν μεγάλη σημασία τα παράκτια και οι ωκεανοί μας. Άρα δεν πρέπει να αλλιεύουμε το, το, το μεγαλύτερα δυνατά ε, πόσο στα υποσά, αλλά να δούμε ποια είναι η αξία για τους πολίτες ε, σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες, τα παράκτια και τους ωκεανούς. Η γραφική παράσταση για τον άξονα 4 και ο συνολικός προϋπολογισμός από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας βλέπω την κατανομία αναχώρα και βλέπω ότι η Ισπανία έχει τη μεγαλύτερη ποσοστή αναλογία του από το συνολικό ποσό που διατίθεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας ενώ η Πολωνία έχει υψηλό ποσοστό ε, και μπορείτε να μας πείτε γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας. Ε, δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο γιατί θα ήθελα να ολοκληρώσετε σε 3-4 λεπτά. Ah, sorry. Je vais répondre en français si vous voulez, je sais pas quoi. Ah, bon, blue. Σε σχέση λοιπόν με την ε, γαλάζια ανάπτυξη, Ήδη εδώ και ορισμένο ε, καιρό είχα ασχοληθεί με αυτή την ε, εργασία και στο Τρινιτάντ και τον Πάκο. Η μελέτη δεν ήταν δική μου και δεν συμφωνώ με τα αριθμητικά στοιχεία, όμως αύριο θα δω κατά πόσο μπορούμε να λάβουμε υπόψη ιδιαίτερα τον ε, τουρισμό. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία στην έκθεση. Ένα 10% διατίθεται στον τουρισμό. Ε, δεν είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο υπολογισμού και χρειάζεται επικαιροποίηση. Γι' αυτό θα μεταβώ αύριο για να το συζητήσουμε ε, δεν συντονίζει τη δραστηριότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ενδιαφέρεται άμεσα. Ε, θα πω για αυτή την εισήγηση σήμερα και θα προσπαθήσουν και οι ίδιοι να δώσουν πιο λεπτομεριακά στοιχεία για τον τουρισμό, για το, τα ταξίδια, φεστιβάλ, κατοικίες και ούτω καθεξής. Εάν ενδιαφέρεστε, μπορώ να αποστείλω στην Επιτροπή Αλίας τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία σε σχέση με τη γαλάζια απασχόληση, δηλαδή να σας δώσω τον συσταλτικό και τον διευρυμένο ε, ορισμό σε σχέση με τα ποσοστά που αφορούν τον ε, τουρισμό. Αλλά πρόκειται για εκτιμήσεις του Μαρτίου του 2014. Μετά θα κάνουμε και προβλέψεις. Ως προς το άλλο ερώτημα... Δεν μπορώ να σας απαντήσω λεπτομερέστερα. με πιο επίκαιρα στοιχεία. Τώρα, σε σχέση γιατί υπάρχει διαφορά μεταξύ του άξονα 4 γενικότερα και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλείας. Ε, ο άξονας 4 βασίζεται στη ζήτηση, δηλαδή εκεί όπου υπάρχει ζήτηση με σημεούλες και... Α, για, για τα flags, δηλαδή σε σχέση με τις... Ε, ε, πρωτοβουλίες που λαμβάνονται ε, με βάση τον άξονα 4. Εάν τώρα η Ισπανία έδειξε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, υπήρξε μεγάλη ζήτηση, δεν σημαίνει ότι θα έπαιρνε ε, όλα τα project γιατί αυτό που ενδιαφέρει είναι η παραγωγή, το marketing παράγουν πάρα πολύ. Η Πολωνία και τα νεότερα κράτη-μέλη έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον διαφοροποίησης για τις περιοχές. Πολλές φορές υπάρχουν επιμέρους προβλήματα, αλλά τους ενδιαφέρει η επιτόπια ανάπτυξη και ο τουρισμός για να προωθήσουν αυτή τη δραστηριότητα όχι μόνο τον τουρισμό, γιατί υπάρχουν και άλλες παράπλευρες επιπτώσεις με βάση ε, εξωτερικούς παράγοντες, άρα υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τον άξονα 4 από την ε, Πολωνία, Ρουμανία και ούτω καθεξής, αλλά και για τους ε, άλλους άξονες που σχετίζονται με την Αλία. Ε, δεν έχω μιλήσει με τις αρχές για τη διάρθρωση αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, παρουσίαση, η οποία και έληξε. Και διακόπτουμε για ένα λεπτό. Ένα λεπτό διακόπτουμε γιατί περιμένει η Επίτροπος. Απλώς θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή στις 20 Φεβρουαρίου ε, ασχολήθηκε, μάλλον έβγαλε μία ανακοίνωση για τον παράκτιο τουρισμό και αυτό σχετίζεται με όσα συζητήσατε εδώ. Υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό και για τον τομέα της αλίας, πολύ περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα για τον ε, παράκτιο τουρισμό και το όλο θέμα συζητήθηκε γιατί ε, οι μελέτες σχετίζονται από το 2010 και μετά σε σχέση με τον θαλάσσιο τουρισμό, δηλαδή το έντρι των τουριστικών δραστηριοτήτων αφορούν τα παράλια, τα και ως προς τον αλλιευτικό τουρισμό που προαναφέρεται. Είναι μορφές ε, τουρισμού που δίνουν πολύ περισσότερα ε, προνόμια σε σχέση με τον παλαιό ε, τουρισμό που λιαζόταν κανείς ε, στον ήλιο. Ωραία, θαυμάσια, σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα συνεχίσουμε την παρουσίαση της Επιτροπής. Συνεχίζουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έκτακτο σημείο της ημερήσία διάταξης. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Επίτροπο στην Επιτροπή μας. Έλεγα την Πέμπτη στην Ολομέλεια ότι κρίμα που δεν ήταν παρούσα η Επίτροπος γιατί ήταν στη Θεσσαλονίκη. Δεν το είπα έτσι με αρνητική χρειά. Ε, έλεγα ότι η ίδια θα στενοχωρηθεί περισσότερο, γιατί εγώ ήθελα να τη συγχαρώ, σπάνια ευκαιρία. Οπότε τώρα έχω την ευκαιρία να τη το πω προσωπικά, συγχαρητήρια, γιατί από ό,τι φαίνεται το αποτέλεσμα μιας μακράς όσο και δύσκολης διαπραγμάτευσης δεν ήταν κακό. Και το λέω γιατί υπάρχει μια καταγγελία, ένα παράπονο στην Επιτροπή μας, ότι δεν είχε εγκαίρως όλα τα στοιχεία στη διάθεσή της για τα ε, όσα διεμήφθησαν η Επίτροπος ήταν δικαιολογημένος απούσα από την Ολομέλεια και προσφέρθηκε να έρθει στην Επιτροπή μας να μας εξηγήσει τι έγινε και βεβαίως όταν λέμε τα ε, αρνητικά θα πρέπει να λέμε και τα θετικά αμέσως. Αμέσως ήρθα σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κανόνισε η Επίτροπος ε, να έρθει σήμερα στην Επιτροπή μας, προσάρμοσε το πρόγραμμά της και την ευχαριστώ ειλικρινά γι' αυτό, γιατί καμιά φορά μπορεί ε, να σας Είχαμε προσάψει κάποια θέματα, τώρα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα πρέπει και δημόσια να το πούμε αυτό που καταφέρατε να έρθετε. Έχουμε λίγο χρόνο, μισή ώρα μόνο, δεν θέλω να μακρηγορήσω, όλοι οι βουλευτές θέλουν να ακούσουν την κυρία Επίτροπο και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, παρακαλώ κυρία Δαμανάκη, έχετε το λόγο και ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και για την ευγενή εισαγωγή. Αφού δεν έχουμε πολύ χρόνο, επιτρέψτε μου να πω στην ουσία του θέματος αμέσως. Να ζητήσω συγγνώμη που δεν είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ήμουν στη Θεσσαλονίκη και συμμετείχα εκεί σε μια διεθνή διάσκεψη κατά της υπεραλίευσης και δεν μπορούσα αυτό να το αναβάλω διότι ήταν εντολή από το Συμβούλιο μας και μάλιστα ομόφωνη να μεταβώ σε αυτή τη ε, διάσκεψη για μια συμφωνία και ήταν δέκα πολύ σημαντικές εκπροσωπήσεις από όλο τον κόσμο που ε, οι δύο αντιπροσωπείες αυτές έχουν υπογράψει αυτή τη διακήρυξη κατά της υπεραλίευσης. Η Ιαπωνία, οι Ηνωμένε Πολιτείε και πολλές αφρικανικές χώρες ήταν παρούσες και τώρα έχουμε αυτή τη δήλωση που εγκρίθηκε ομόφωνα από τα δικά μας κρατημέλη συν τους φίλους μας και εταίρους. Λοιπόν, για τη συμφωνία την ίδια να σας δώσω μια σύντομη παρουσίαση των όσων συμφωνήσαμε και ίσως ακολουθήσει και συζήτηση. Νομίζω ότι είναι καλή τελικά αυτή η συμφωνία και θα ήθελα να το πω με τρόπο πάρα πολύ ξεκάθαρο ευθύ εξ αρχής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ ε, και δημόσια ε, τις ομάδες μας ε, για τις καλές υπηρεσίες. Γιατί είναι καλή η συμφωνία. Διότι μετά τη συμφωνία αυτή θα τερματιστεί μια χαόδης κατάσταση που επικρατούσε στο Βόρειο Ατλαντικό σχετικά με τα θέματα σκόμβρου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και πολλές οι συγκρούσεις. Κάποιες εφημερίδες έγραψαν και μέχρι για τον πόλεμο του σκουμπριού. Και μέχρι κάποιο βαθμό αυτό είναι γεγονός. Υπήρξαν τεράστιες συγκρούσεις ε, από τις ε, παραθαλάσσιες χώρες ε, με εμά, την Νορβηγία, την Ισλανδία, η νήσι Φαρόε, οι πάντες ήταν κατά των πάντων. Νομίζω τώρα έχει τερματιστεί αυτό το χάος, τεράστιο χάος επικρατούσε εκεί. Λοιπόν, ε, έχουμε πλέον μια ε, συμφωνία πενταετούς διάρκειας. Ε, το πρώτο έτος θα υπάρξει μια λύση ad hoc μόνο για τη χρονιά αυτή. Θα το χαρακτήριζα μεταβατικό αυτό για να πιστούν οι πάντες για τη συμφωνία αυτή. Από το επόμενο έτος, το δεύτερο, όλοι ε, θα δεσμεύονται να αλλιεύουν ε, σε βιώσιμη βάση. Για την επόμενη τετραετία, δηλαδή μετά τη μεταβατική χρονιά, θα είναι βιώσιμη αλλία και αϊφόρος και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το μέλλον. Δεύτερον, επαναφέραμε και αποκαταστήσαμε και πάλι τις σχέσεις μας με τις νήσους Φαρόε είναι πολύ σημαντικό αυτό, όχι μόνο για πολιτικού λόγου, αλλά και για τα δικά μα κράτη-μέλη, διότι μπορεί να γνωρίζετε, σίγουρα γνωρίζετε, είμαι βέβαια, ότι πολλά από τα δικά μα κράτη-μέλη έχουν ε, αλλιευτικά συμφέροντα και έχουμε σκάφη που δεν αλλιεύουν σκουμπρί, αλλά άλλα είδη, ενώ και γύρω στις νήσους Φαρόε και πολλά σκάφη δικά μας ενδιαφέρονται και έχουν συμφέροντα εκεί οπότε αποκαταστήσαμε τις καλές μας σχέσεις και μπορούμε και πάλι να ψαρεύουμε στα νερά τους. Ε, τρίτον, συμφωνήσαμε με την Νορβηγία διμερός όπως μπορείτε να καταλάβετε η Νορβηγία είναι ένας εταίρος ε, ιδιαίτερα σημαντικός, ίσως ο σημαντικότερος μετά τα κράτη-μέλη μας ε, και ε, γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι και πολλά κράτη-μέλη έχουν ε, μεγάλο ενδιαφέρον επιδείξει να αλλιεύουν εκεί και είμαι σε θέση να σας ανακοινώσω ότι από χτες νομίζω ήδη έχουν μεταβεί εκεί τα σκάφη μας σε νορβηγικά ε, ύδατα και ψαρεύουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τα σκάφη, είναι και πολλές θέσεις εργασίας σήμερα που συνδέονται με αυτό. Δηλαδή εξασφαλίσαμε να μην κινδυνεύουν θέσεις εργασίας. Έχουμε τώρα μία δέσμη, ένα πακέτο, όχι μόνο για το σκουμπρί επαναλαμβάνω, αλλά και μια συμφωνία για τα υπόλοιπα ε, πλήρη ε, και με την Νορβηγία. Για όλα τα αποθέματα και τα είδη ε, που έχουμε κοινή συμφωνία για αυτά. Αυτή είναι η βασική λόγη που νομίζω εγώ ότι είναι καλή και η συμφωνία. Η σταθερότητα, η βιωσιμότητα, καλές σχέσεις με την Νορβηγία και τις νήσους Φαρόε, αλλά ε, μπορούμε ε, και ε, για άλλα είδη να ψαρεύουμε. Μερικές λεπτομέρειες τώρα για την ίδια τη συμφωνία. Είναι πενταετούς διάρκειες, είπαμε. Συμφωνήσαμε για ένα αλλιεύμα για το 2014 1,24 εκατομμύρια τόνους που είναι πέραν της επιστημονικής συμβολής έχουμε αυξήσει το συνολικό επιτρεπτό αλλιεύμα για να μπορέσουν όλοι να συμφωνήσουν και θα εξηγήσω στη συνέχεια και θα σας πω για ποιο λόγο και πόσο. Τα μερίδια που έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη είναι ακριβώς τα ίδια με εκείνα του παρελθόντος. Δηλαδή 49% για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 22% η Νορβηγία και 12,6% η νήσι Φαρόε. Έχουν συμφωνήσει τα μέρη επίσης να επανέλθουν στη σχετική κατανομή που είχαμε μέχρι το 2018. Δεν έγινε καμία παραχώρηση στην Ορβηγία για το μερίδιό της. Από το σονελικό επιτρεπτό ε, αλίευμα έχουμε αφήσει στην άκρη 15,6% επαναλαμβάνω 15,6% και αυτό αναλογεί στην Ισλανδία εάν θέλουν να προσχωρήσουν και οι Ισλανδοί και νομίζω ότι αυτό ε, ισχύει και για τη Γρυλανδία ε, που είναι η αλία της ε, και το αλλιευτικό πεδίο εκεί πειραματικό. Αυτό το 15,6% είναι ένα μερίδιο που αναλογεί στις προσδοκίες όλων, στις μακρές και επίπονες διαπραγματεύσεις. Πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ καλό αυτό το μερίδιο και επιτρέπει στην Ισλανδία να προσυπογράψει τη συμφωνία. Έχουμε τώρα την εξή και μόνη ανησυχία για τη Γρυλανδία. Ξαφνικά η Γρυλανδία στο παραπέντε της υπογραφής της συμφωνίας, γιατί μάλλον το, έμαθε, εμφανίστηκε με μία ποσόστοση μόνο μερή και μεγάλη, 100.000 τόνους, 100.000 τόνους, που μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι παρά ε, της πειραματικής αλίας. Ε, συμφωνήσαμε λοιπόν μαζί τους αλλά δεν... Έχουμε μια συμφωνία μαζί του, αλλά δεν προχώρησε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τη Γρυλανδία για να δούμε πώ θα εξελιχθεί η κατάσταση. Μπορώ να σα πω όμω πολύ ειλικρινά ότι τώρα που έχουμε συμφωνήσει με του υπολείπου και είναι τετελεσμένη η συμφωνία, ε, προσωπικά φρονώ ότι θα είναι πιο εύκολο να συμφωνήσουμε και με τη Γρυλανδία. Είναι προσωπική μου άποψη αυτή. Και πιστεύω ότι ήταν μάλλον αντίδραση τη Γρυλανδία θεωρώντας και πιστεύοντας ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία ε, ε, οπότε θα γίνει μια κούρσα, ένας αγώνας, ο καθένας θα αλλιεύει όσες ποσότητες θέλει και ό,τι θέλει. Για το μέγιστο επιτρεπτό αλλιεύμα, όπως σας είπα, αυξήθηκε ε, πέραν της επιστημονικής συμβουλής που ήταν περίπου 900.000 τόνοι, αυτό που συμβουλεύουν οι επιστήμονες. Εμείς αυτό το υπερεύημεν και πήγαμε στο 1,24. Για ποιο λόγο. Μόνο για ένα έτος δεν θα πειράξει το απόθεμα, διότι... Έχουμε πληροφορίες νέες από τους επιστήμονες πριν από δύο εβδομάδες οι επιστήμονες του ISIS έχουν αναθεωρήσει τις μεθόδους και μας ενημέρωσαν ότι το απόθεμα υπολογίζεται στους 3 με 6 εκατομμύρια τόνους. Επαναλαμβάνω, μεταξύ 3 και 6 εκατομμυρίων τόνων. Σύμφωνα με ε, τις νέες ε, εκτιμήσεις και υπολογισμούς θα διπλαδιασιαστεί. Βεβαίως δεν ήμασταν σε θέση να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα επιστημονικά δεδομένα. Θέλουμε να το συζητήσουμε με την ISIS σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Αλλά δεδομένων αυτών των στοιχείων, δεν λέω ότι είναι απόλυτη αλήθεια, Καταλαβαίνουμε ότι είναι και μεγάλη η ψαλίδα από 3 σε 6 εκατομμύρια τόνους. Αλλά συμφωνούν όλοι, ε, είναι γενική συμφωνία, όλοι οι επιστήμονες συμφωνούν, επαναλαμβάνω, ότι είναι σε καλή κατάσταση τα αποθέματα με τάση αυξανόμενη. Δηλαδή έχουμε 100% παραπάνω από την επιφυλακτική και προσεκτική συμβουλή που μας είχαν δώσει οι επιστήμονες. Νομίζω ότι μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι για το επόμενο έτος μπορούμε να αυξήσουμε την ποσόστοση. Επίσης θα ήθελα να πω ότι έχουμε αρχίσει συζητήσεις με τις νήσους Φαρόε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τα υπόλοιπα αποθέματα και ήδη. Θα θυμάστε ότι έχουμε ήδη επιβάλει κυρώσεις στις νήσους Φαρόε για τη Ρέγκα Και είναι σημαντικό αυτό που κάναμε, διότι τα σκάφη των νήσων Φαρόε θα έρχονται στα δικά μας ύδατα να ψαρεύουν ε, σκουμπρί και δεν θα ε, έχουν ε, παράπλευρα ε, αλλιεύματα ε, ρέγγας. Και ε, θα πρέπει σε παρόμοια επίπεδα να παραμείνει του 13 η ρέγγα. Και σας υπόσχομαι ότι πριν λήξει η θητεία μου με τρόπο ειρηνικό θα συμφωνήσω για αυτό το θέμα με τις Νησφαρόε χωρίς να κινδυνεύει το είδος. Λοιπόν, έχουμε συμφωνήσει, τα τρία μέρη είναι ε, ανοιχτό γιατί έχουμε εξασφαλίσει και μερίδιο για την ε, Ισλανδία όταν θελήσει και με τη Γρυλανδία είμαστε σε επαφή για να μπορέσουμε να το λύσουμε και το ίδιο ισχύει για τις νήσους Φαρό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την ε, Επίτροπο. Αρκετοί έχουν ζητήσει το λόγο. Επτά θέλουν το λόγο. οι διερμηνείς θα μας διαθέσουν λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά όχι περισσότερο. Δεν θα ήθελα να παρέμβετε περισσότερο από δύο λεπτά ο καθένας, έτσι ώστε η Επίτροπος να μπορέσει να απαντήσει. Ο Αντιπρόεδρος Στίβενσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ την Επίτροπο που προσήλθε εδώ για να μας δώσει ε, τις δέουσες πληροφορίες. Θα ήθελα να σας συγχαρώ, ε, εσάς και τον Τζον Spencer διότι αντέξατε τρία χρόνια ε, μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, συνεπώς επιτύχατε, αλλά το πρόβλημα είναι ότι η συμβουλή του ISIS μιλάει για ένα φάσμα 3 με 6 εκατομμύρια τόνους. Όταν αρχίσαμε αυτό τον πόλεμο, ε, για το σκουμπρί είχαμε ε, ένα ανώτατο επιτρεπτό αλίευμα 540.000 τόνων και φαίνεται ε, ότι έχει διπλασιαστεί τουλάχιστον το ε, απόθεμα σε σχέση με το αρχικό ανώτατο επιτρεπτό αλίευμα για το ε, σκουμπρί. Και βεβαίως υπάρχει και ο γόνος, ο οποίος είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Άρα το αλίευμα είναι υψηλότερο. Τι θα συμβεί και τι θα συμβεί αν ε, φτάσουμε ξανά στις 540.000 ε, τόνους, διότι μιλάμε για ένα 15,6% ε, στην Ισλανδία και τη Ρωσία, 12,6% στις Φερόες νήσους και 100.000 ε, τόνους ε, για τη Γρυλανδία. Δηλαδή μας μένουν 150.000 τόνοι για τη Νορβηγία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό πραγματικά με ανησυχεί. Γιατί όλοι οι αλλοί θα λένε ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά, αλλά σε πέντε χρόνια δεν θα είναι και τόσο ευτυχής εάν φτάσουμε στο σημείο που ξεκινήσαμε από το σημείο εκκίνησης δηλαδή. Στο μεταξύ όμως θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ με εκπληση διότι η Ισλανδία δεν ε, άδραξε αυτή την ευκαιρία, άρα χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα που έχετε για να επιβάλλετε σκληρές κυρώσεις. Όχι μόνο για το σκουμπρί, αλλά και όλα τα συναφή αποθέματα ε, στα ύδατα αυτά. Άρα να φτάσουμε σε συνολική συμφωνία με τις κυρώσεις. Δεν θέλω να υπερβείτε τα 12 λεπτά, ο κύριος ε, Βαλέσα και μετά Ντότσα. Ίσως χρειαστώ 2,5 λεπτά. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε κυρία πίτροπε. Δύο ερωτήσεις. Βλέπουμε μία κίνηση ορισμένων αποθεμάτων περισσότερο προς το βορρά. Στην περίπτωση της Γρυλανδίας αυτό σημαίνει νέες δυνατότητες και ευκαιρίες. Η Γρυλανδία ίσως να μην μπορέσει να χρησιμοποιήσει ε, τη δυνατότητα αυτό του αποθέματος. Και αυτό σχετίζεται και με το σκουμπρί. Το 2013 και κατά προγενέστερα έτη η δραστηριότητα των Κινέζων και των Ρώσων στη Γρυλανδία έχει αυξηθεί ραγδαία. Οι οικονομικοί τους φορείς είναι παρόντες σε αυτά τα ε, συμπεριλαμβάνοντας και το, την εταιρεία Lafayette που ασχολείται ε, περισσότερο με τις αλλιότρατες, αλλιεύοντας 15.500 ε, τόνους ημερησίως. Αυτό, που έχει σημασία, αυτό έχει μεγάλη σημασία στρατηγικά. Επίσης μία μόνιμη, υπήρχε μία μόνιμη συμφωνία με τη Γρυλανδία που επιτρέπει νέες αλλιεύσεις θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και για το σκουμπρί κατά βιώσιμο τρόπο. Εάν αποτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να φτάσει σε μια τέτοια συμφωνία με τη Γρυλανδία, δηλαδή μια φόρμουλα καθαρού κέρδους, τότε θα μπορέσει να υπάρξει εκμετάλλευση παρόμοια εκμετάλλευση και σε άλλους τομείς και ίσως αυτοί οι πόροι, αυτούς τους πόρους τους αδράξουν οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Αυτό θα ήταν ολέθριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω λοιπόν να, γίν, ε, να λάβουμε υπόψη ότι ορισμένες από τις παραχωρήσεις της Επιτρόπου δεν θα πρέπει να παραμείνουν. Αυτό το θεωρώ στρατηγικό λάθος. Άρα θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα υποστηρίξετε τη ε, μέσα στα πλαίσια αυτής της νέας βιώσιμης δραστηριότητας και πώς μπορείτε να ενισχύσετε το ρόλο της Γρυλανδίας στο Βόρειο Ατλαντικό. Με την ευκαιρία αυτή, επειδή δεν ήσασταν παρούσα την προηγούμενη εβδομάδα, ε, ασχοληθήκαμε και με το Χάλιμπατ, στην βόρεια, στα βόρεια ύδατα. Ο κανονισμός J87 του 2001 ε, λαμβάνουμε υπόψη τη, το περιορισμό κατά 50% του κόκκινου μπακαλιάρου στις ε, Φερόες και στη Γρυλανδία. Τι έκανε η Επιτροπή για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα και ε, διαφορετικά υπάρχει ένας μηχανισμός αντιστάθμισης για τους οικονομικούς φορείς που αυτή τη στιγμή ε, υφίστανται μία διάκριση με βάση τις ε, οικονομικές συνέπειες. Ευχαριστούμε κύριε πολύ, πολύ κύριε ε, Βαλέσα δεν μπορούν να είναι τόσο σχηνοτενείς ε, οι ερωτήσεις. Dodge. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και γεια σας κύριε Επιτρόπε. Τρία σημεία. Ο κύριος Στίβενσον βασικά με κάλυψε. Φαίνεται πως υποχρεωθήκαμε να βρεθούμε σε μια θέση. Πριν τρία χρόνια ξεκινήσαμε να συζητούμε για το σκούμπρι και τότε η ποσόστηση ήταν 540.000 και τώρα έχουμε φτάσει στα 6 εκατομμύρια και η ψαλίδα είναι τεράστια. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά από ε, ε την επιστημονικές ε, συμβουλές που λάβαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ελπίζω, ελπίζω πραγματικά να μην έχουν πειραχτεί αυτά τα στοιχεία που μας έδωσε το ISIS προκειμένου να επιτύχουμε πολιτική συμφωνία. Επίσης, στο θέμα του κόνου που έθεσε ο κ. Στρούν. Εάν λάβουμε υπόψη μας την ε, συμφωνία αυτή τη στιγμή, είναι αναποφευκτό όταν μειωθεί το αλληλευτικό απόθεμα, τα ποσοστά θα παραμείνουν και θα έχει αυτό ως αποτέλεσμα οι αλληλείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να αλλιεύουν λιγότερο. Επίσης, το ΤΑΚ αυξάνεται πολύ σημαντικά στη τη χρονιά αυτή και θα ήθελα να γνωρίζω την άποψή σας ποιες επιπτώσεις θα έχει αυτό για την τιμή του σκουμπριού και αν αυτό δεν θα επηρεάσει δυσμενώς και την, τον κλάδο. Η κυρία Παθαθάου. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε που επισκεφθήκατε την Επιτροπή μας με αυτά τα καλά νέα, αλλά τα γνωρίζαμε ήδη. Γι' αυτό εγώ θα εστιάσω περισσότερο στις ανησυχίες που έχω για την ε, συμφωνία. Το θέμα της Γρυλανδίας ήδη αναφέρθηκε, εγώ όμως θα αναφερθώ στην Ισλανδία. Είπατε ότι η πόρτα είναι ανοιχτή, αλλά εκείνοι δεν θέλουν να την περάσουν. Δεν θέλουν να συμφωνήσουν. Όμως μια τριμερή συμφωνία δεν επαρκεί Ιδιαίτερα γνωρίζοντας την σημασία και την ε, έντονη δραστηριότητα που αναπτύσσει η Ισλανδία στην, περιοχή. Επομένως με ανησυχεί πραγματικά το γεγονός ότι δεν συνυπέγραψαν τη συμφωνία και θα ήθελα να μου πείτε τι, πρόκειται, τι πιστεύετε ότι πρόκειται να συμβεί βράχη πρόθεσμα στο, στο, στο μέλλον τώρα κοντά. Δεύτερο σημείο. Ακούσαμε πολλούς αριθμούς, πολλά αριθμητικά στοιχεία. Όμως θα ήθελα να το μηνύσω ότι ο ίδιος ο κλάδος της αλίας λέει ότι η ηχθειοκαλλιέργεια ότι μάλλον με τη συμφωνία που έγινε ότι αναμένουν να μειωθεί η αλία κατά 20% και αυτό το λέει ο ίδιος ο κλάδος. Με άλλα λόγια ο ίδιος ο κλάδος μας λέει ότι δεν θα αποκομίσει ωφέλη από αυτή τη συμφωνία. Εκείνοι που θα αποκομίσουν ωφέλη, εκείνοι που θα αποζημιωθούν, εκείνοι που θα αποκομίσουν ωφέλη ουσιαστικά είναι κυρίως εκείνοι που δεν ε, τηρούσαν τους παλαιότερους κανόνες, δηλαδή τα είναι Στην πραγματικότητα υποστηρίζουμε και βοηθάμε εκείνους που παραβίαζαν τους κανόνες. Εκείνοι που τους παραβίαζαν, όπως για παράδειγμα η Φερόε, δεν αναγκάζονται, δεν εξαναγκάζονται να πληρώσουν για αυτές τις παραβιάσεις και αντιθέτως τους ε, υποστηρίζουμε κι άλλο. Ευχαριστώ κύριε Πατρά. Ο κύριος ε, Γκάλαχερ, ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπε ε, ο κύριος Στίβενσον, η κυρία Τότς. την περασμένη Πέμπτη στην Ολομέλεια μάθαμε τα νέα για τη συμφωνία, τη στιγμή που επρόκειτο να ψηφίσουμε. Ε, μετά από λίγες ώρες ουσιαστικά. Μου είπε η γραμματεία ότι ενημερώθηκε από τον τύπο για τη συμφωνία. Θα προτιμούσαμε να τα μάθουμε από πρώτο χέρι και όχι από δημοσιεύματα. Μήπως θα μπορούσατε κύριε Επίτροπε αυτό να το επιβεβαιώσετε, να το διαψεύσετε. Και τέλος μιλήσατε για μια συμφωνία ε, με τις νήσους ε, Φερόε για το σκουμπρί για τα παράπλευρα αλλιεύματα ότι ήταν με το πιστόλι στο πρόταφο. Μα όχι, συγγνώμη, μιλήσατε για ειρηνική συμφωνία ότι θέλετε. Ε, ε μπορεί να δείξουν απροθυμία να συμφωνήσουν ειρηνικά. Τι θα κάνετε, ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Γκάλεχερ, ε, ήταν ο κύριος Άγνου. Ευχαριστώ, συμφωνώ με τον κύριο Άγνου. Μέχρι τις 9 και 40 συζητούσαμε και την ίδια μέρα, την ίδια μέρα ε, δεν πήραμε τη συμφωνία ε, από εσά. Ε, και είναι κρίμα και είναι πολύ σημαντική η Επιτροπή μας. Μας έχετε αγνοήσει πλήρως και απολύτως. Σήμερα το πρωί τόσο αργά μας είπανε να πάμε στον Περλεμόντ να πάω αντίγραφο. Κυρία Επίτροπε, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν ξέρω ποιο θέλει. Εσεί είστε πολιτικά υπεύθυνοι και επικεφαλή και αυτό αποτελεί ύβρι και προ εμένα και προ υπολείπου. Ωραία ε, να ε, συγχαίρουμε τους ανθρώπους πιστεύετε στην αηφορία, πιστεύετε στη βιωσιμότητα και πώς το λύνετε από 100.000 τόνους φτάσατε στα 1,24 εκατομμύρια. Συμφωνώ και με την κυρία Τότς και τον κύριο Στίβενσον. Από 57 έχουν αυξηθεί πάνω από 100 στην Ιρλανδία και ε, θα μειωθεί η ε, θέση μας στην αγορά. Οι μεγάλοι νικητές εδώ δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Φαρό και η Ισλανδία που όλα αυτά τα χρόνια ε, έκαναν και είχαν αυτή την τακτική που είχαν. Γιατί να τους δώσουμε 15% δίνουμε στην Ισλανδία, τι συμφέρον έχει να ενταχθεί η Ισλανδία. Τον Ιούλιο μας υποσχεθήκατε εδώ στην Επιτροπή ότι θα αρχίσετε τη διαδικασία για τις κυρώσεις. Εδώ σήμερα δεν βλέπουμε πουθενά αναφορά σε κυρώσεις. Για το 2015 λέγεται ε, θα γίνει σιγά σιγά βιώσιμο. Ε, γιατί το λέτε και πώς το λέτε, το ΤΑΚ ποιο θα είναι το 15, το 16, το 17, πώς μπορείτε να το προβλέψετε. Μπορεί να ήταν καλή συμφωνία για ορισμένες χώρες, αλλά μπορώ να σας εγγυηθώ ότι αν δεν καταρρεύσει θα μειωθεί η τιμή, εκτός εάν ε, λάβετε κάποια δράση έναντι της Ισλανδίας. Και την άλλη εβδομάδα θα πάω και θα τους τα πω κιόλας. Αλλιώς θα καταρρεύσουν. Και φταίει το γραφείο σας που δεν μας έχει δώσει ενημέρωση. Για ποιο λόγο να μην τα γνωρίζουμε εμείς στην Επιτροπή μας. Έχουμε δικές μας απόψεις και τις λέγουμε. Και δεν υποκλεινόμαστε κάθε φορά, ούτε βγάζουμε το καπέλο στην Επιτροπή και στις υπηρεσίες της Επιτρόπου. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόμας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την Επίτροπο για αυτές τις διασαφήσεις πολύ γρήγορα γιατί οι άλλοι συνάδελφοι υπέβαλαν τις καλές ερωτήσεις. Ε, συμφωνώ με τον κύριο Γκάλαχερ για τις ε, ε, ε κυρώσεις έναντι της Ισλανδίας και της Γρυλανδίας και τις ανησυχίες που εκφράσαμε για τα μελλοντικά χρόνια ως προς τις ποσοστώσεις και το θέμα των τιμών. Ως προς την Νορβηγία, μπορείτε να μας πείτε τώρα ή λίγο αργότερα πόσα σκάφη ενέχονται σε αυτή την ε, αλίευση στα παράκτηρα της ε, Νορβηγίας. Η ε, Επίτροπος μπορεί να απαντήσει a few explanations about the procedure. Uh, Ορισμένες διευκρινήσεις. Πρώτα απ' όλα, αμέσως μετά την συμφωνία έδωσα την εντολή το επιτελείο μου να ενημερώσει τον κύριο Μάτου και εσάς τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, για το γεγονός αυτό ε, της συμφωνίας. Επίσης ζητήθηκε, ζήτησα να σας δοθεί αμέσως ένα αντίγραφο ε, ζητώ συγγνώμη αν αυτό δεν συνέβη, αν δεν το έκανε η η, οι υπηρεσίε τι οποίε επιβλέπω. Πάντω, εάν συνέβη αυτό, θα το εξετάσω. Πάντω, ε, κατά την άποψή μου, ενημερωθήκατε. Δεν το μάθατε από τι εφημερίδε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Να καταλάβω. Το προηγούμενο βράδυ, αμέσω μόλι συμφωνήσαμε, αμέσω μόλι υπογράψαμε, εγώ επικοινώνησα τον κύριο, με τον κύριο Μάτου και τον κύριο Γκάλαχερ και του ενημέρωσα. Την επόμενη μέρα ήσασταν στο κοινοβούλιο και βεβαίω το, το, κείμενο δεν υπήρχε ακόμα εκεί στο κοινοβούλιο. Ε, ωστόσο ο πρόεδρος της ε, Επιτροπής της κοινοβουλευτική μου λέει ότι το κείμενο το λάβατε μόλις σήμερα. Αυτό είναι λάθος. Θα μάθω τι έγινε, θα μάθω γιατί δεν ε, λάβατε αμέσως το κείμενο, γιατί δεν υπήρχε και τίποτα να κρύψουμε ε, Θεού. Πιστεύετε τώρα εδώ ότι το κάναμε εσκεμένα. Λάθος μας. Είμαι απολύτως πεπισμένη, κύριε Κάλαχερ, ότι έχουμε πολύ καλές Επικοινωνίε Πολύ καλή μάλλον επικοινωνία με τον κλάδο. Επομένως δεν θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα όταν δίνουμε κάτι στους προσώπου του κλάδου να το μοιράζομαι και μαζί σας. Ε, είναι δυνατόν τώρα να υπάρχει κάποιο ένα κείμενο το οποίο δεν θέλω να μοιραστώ με το κοινοβούλιο και να το δίνω στους, στους, ε, του κλάδου. Ήθελα να είμαι απολύτως σαφής από αυτό. Λοιπόν, αυτό για το ζήτημα της διαδικασίας. Αλλά το θέμα είναι το θέμα ουσίας, όχι τόσο διαδικασίας. Λοιπόν, στο μέλλον ε, σας εγγυώμαι οτιδήποτε συμφωνείτε θα το λαμβάνετε αμέσως, έχετε κάθε δικαίωμα, ε, συμφωνώ μαζί σας ότι ήταν λάθος που δεν το λάβατε, θα το φροντίσω. Λοιπόν, για το ζήτημα των επιστημονικών στοιχείων. Πρέπει να τα σέβομαι. Δεν μπορώ να υπονομεύσω ή να πω ε, εκ των προτέρων ότι αυτά τα επιστημονικά στοιχεία είναι λάθος, όπως ορισμένοι από εσά τους βουλευτές το κάνουν. Γιατί εάν ξεκινήσει μια τέτοια ε, συζήτηση ότι τα επιστημονικά στοιχεία είναι λάθος υπηραγμένα, δεν έχουμε καμία βάση συζήτησης. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να διαρευνήσω και να μάθω με ποιον τρόπο οι επιστήμονες έχουν καταλήξει τα συμπεράσματα που μας δίνουν. Πριν την συζήτηση, πριν από τη συζήτηση για τη συμφωνία φέτος, οι επιστήμονες που συμβουλεύόμαστε μας είπαν πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι το απόθεμα αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό του ζητήσαμε με προτάσει και οι προτάσει που μαθαίνονταν ήταν εκείνε. Ήταν ένα τάκ ε, τη τάξη των 900.000 τόνων. Τώρα λένε ότι ακριβώ λόγω αυτή τη μεγάλη αύξηση του, ε, του αποθέματο θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα πέρα-πέρα. 3 6 εκατομμύρια. Αλλά για αυτό ακόμα δεν έχουμε απόδειξη επιστημονικά στοιχεία. Επομένως τα 3 6 εκατομμύρια που σας είπα είναι απλώς υποθετικά δεν είναι κάτι το οποίο αποφασίσαμε. Είναι μια πιθανότητα. Εάν συνεχίσει να αυξάνεται το ελευτικό απόθεμα, κάτι τέτοιο προβλέπουμε για την επόμενη χρονιά. Δεν είναι όμως ένα νούμερο το οποίο σα το δίνω ως ε, συμφωνημένο ή αποφασισμένο τα 3-6 εκατομμύρια. Το αποφασισμένο είναι 900.000 τόνοι. Και για του χρόνου είπαμε 1,2 ε, εκατομμύρια θα προτείνουμε και αν μετά συμφωνήσουν όλοι θα προχωρήσουμε. Ακολουθούμε λοιπόν τα επιστημονικά στοιχεία. Δεν μπορώ να προβλέψω ποια θα είναι η ποσόστοση το 2015 το 2016, γιατί θα πρέπει πρώτα να λάβουμε τα επιστημονικά στοιχεία. Αυτό που πάντως συμφωνήσαμε και καταφέραμε να συμφωνήσουμε είναι ότι όλοι συμφώνησαν ότι θα ακολουθήσουμε την επιστημονική ε, στι των επιστημόνων. Δηλαδή ό,τι πουν του χρόνου οι επιστήμονε, θα το ακολουθήσουμε. Αυτή είναι η συμφωνία. Μην υπάρχουν παρανοήσεις. Τώρα, σε σχέση με τα ποσοστά. Την κατανομή των ποσοστών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νορβηγία έχει τα ίδια ποσοστά. Επίσης, το νορβηγικό ποσοστό είναι ακριβώς το ίδιο με το προηγούμενο. Επομένως, γιατί σας δημιουργεί ανησυχία. Φυσικά, εάν το απόθεμα αρχίσει να μειώνεται και υπάρχουν προβλήματα και μειωθεί και η ποσότητα, έτσι θα γίνει. Αλλά τα ποσοστά παραμένουν. Μειώνεται το συνολικό ποσό, η ποσόστοση, αλλά η κατανομή των ποσοστών δεν αλλάζει. Και αυτό θεωρώ μάλιστα ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματά μα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό ε, δημιουργεί προβλήματα. Αντιθέτω, ο κλάδο ήταν ενθουσιασμένο από αυτό. Ήταν ε, μάλιστα οι αντιδράσεις του ακόμα πιο θετικέ από ό,τι περίμενα για να είμαι ειλικρινή. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν είναι κάτι το οποίο συμφωνήσαμε για του χρόνου. Δεν είναι ότι είπαμε ότι αν πάμε σε τάκ 1,2 εκατομμύρια τότε θα είναι τα ποσοστά έτσι. Τα ποσοστά είναι αυτά και θα συνεχίσουν να είναι. Και μάλιστα το είχαμε συζητήσει κύριε Γκάλαχερ γιατί έρχεστε και μου παραπονείστε τώρα. Πραγματικά θέλω να το καταλάβω. Ακριβώς τα ίδια ποσοστά και ακριβώς η ίδια κατανομή ποσοστών θα έχουμε. Τι πρόβλημα παρουσιάστηκε. Ναι, εάν το επόθεμα αυξηθεί ε, το ποσοστό αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο ε, σε μεγαλύτερη ψαριά. Εάν το απόθεμα μειωθεί, αντιστοίχω θα μειωθούν και τα αλλιεύματα. Η εξαίρεση είναι μόνο για, του, για φέτος. Φέτος ξεπεράσαμε τις επιστημονικές συστάσεις απλώς και μόνο για να επιτύχουμε τη συμφωνία. Τώρα που την επιτύχαμε τη συμφωνία έχετε δίκιο είναι και τίθεται το θέμα τι θα κάνουμε με του υπόλοιπου. Και εδώ συμφωνώ με τι ανησυχίε που εκφράζεται. Ε, ε, τι συμμεριζόμαστε κι εμεί. Γι' αυτό προσπαθούμε να δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε τη Γρυλανδία και την Ισλανδία. Πάντω, σε κάθε περίπτωση, έχουμε αφήσει στην άκρη ένα σημαντικό ποσοστό. Επομένω, εάν η Ισλανδία συνεχίσει να αλλιεύει όπως ήθελε 12-13% τότε παραμένει η συνολική αλλία σε ασφαλές επίπεδο. Τώρα το ζήτημα των μέτρων, των κυρώσεων που θα αναλάβουμε εναντίον της Γρυλανδίας. Θα δούμε. Θα δούμε. Πρέπει να συζητήσω πρώτα μαζί τους, θα τους καλέσουμε, θα παραστώ θα, θα επισκεφτώ μάλλον την Ιρλανδία, θα συζητήσουμε για το ζήτημα της, πειραμα, πειραματικής αλίας, αλλά τώρα μην ξεχνάτε ότι είμαστε τρεις, θα πάμε μαζί με τους Νορβηγούς, μαζί με τους Ιρλανδούς. Επίσης, επολύτως ειλικρινά να σας πω και νομίζω καταλαβαίνετε γιατί δεν ξέρω τι θα κάνουμε με τη Ρωσία αλλά πάντως η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα είναι καλύτερη από την προηγούμενη, γιατί παλιότερα τι είχε συμβεί, η Ρωσία και η Νορβηγία είχαν μια διμερή συμφωνία. Επομένως, εάν δεν είχαμε καταφέρει να συμφωνήσουμε με τους Νορβηγούς, ε, θα ήμασταν σε χειρότερη μοίρα. Νομίζω όλοι καταλαβαίνετε. Άρα, παρά το γεγονό ότι είμαστε τρει, είμαστε σε καλύτερη θέση. Ναι, για τη Ρωσία, για την Νορβηγία και την Ισλανδία Υπάρχουν ανησυχίε, αλλά είμαστε σε ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση σήμερα από ό,τι στο παρελθόν. Δεν μπορώ να σα απαντήσω τώρα αυτή τη στιγμή ε, πώ εκατοντάδε πάντω είναι πόσα σκάφη τη Νορβηγία αλλιεύουν στι ε, περιοχέ αυτέ, τα είδα αυτά. Πάντω θα το ζητήσω από τι υπηρεσίε μου να σα ενημερώσουν για τον ακριβή αριθμό. Πάντω η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη, λίγο περίπλοκη εκεί, γιατί θεωρεί η Νορβηγία ότι είναι κυριαρχικό του δικαίωμα να αλλιεύει στα εθνικά τη ύδατα ε, είναι ένα θέμα στο οποίο δεν θέλω να λάβω τώρα μια απόφαση. Πρέπει να συνεργαστούμε και να το συζητήσουμε μαζί μα και να καταλήξουμε στο ποια θα είναι η θέση. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και ε, αντικρουόμενε απόψει μεταξύ των ιδίων των κρατών μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό προσπαθώ να είμαι προσεκτική εδώ. Και τελευταίο θέμα για το μέλλον. Θα συζητήσουμε με τους εκπροσώπους του κλάδου, θα επισκεφθούμε τη Γρυλανδία θα συζητήσουμε και με την Ισλανδία. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει εάν με από όλα αυτά η Ισλανδία δεν συμμετάσχει στη συμφωνία. Θα εξετάσουμε όλα τα πιθανά μέτρα που μπορούμε να λάβουμε και να αντιδράσουμε με βάση και συμπεριλαμβανομένο των νομικών εργαλείων που έχουμε στα χέρια μας. Με άλλα λόγια όμως δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή τι κυρώσεις ή με ποιον τρόπο θα κινηθούμε εναντίον τους. Πολλά πράγματα είναι ασαφή πρέπει να δούμε πώς θα αναθεωρήσει και τις υποστημικές συστάσεις του ISIS, να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει με το απόθεμα, το οποίο κινείται προς τα, βόρεια, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν έχουμε συγκεκριμένα ε, στοιχεία να γνωρίζουμε ακριβώς τις κινήσεις του. Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες πριν να λάβουμε αποφάσεις, έχοντας τα επιστημονικά στοιχεία στα χέρια μας. Καταλαβαίνω λοιπόν τη ανησυχία μας, αυτό θα ήθελα να πω συμπερασματικά, αλλά και εμείς τα ίδια πράγματα μας ανησυχούν. Το ζήτημα της Ισλανδίας, το ζήτημα της Γρυλανδίας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και θα βρισκόμαστε σε επικοινωνία. Τώρα, αν εσείς έχετε κάποια καλή ιδέα με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τους Γρυλανδούς, ευχαρίστω. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχω λάβει κάποια πρόταση. Πολύ θα ήθελα να δω πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Όλα είναι ανοιχτά, όλες οι πιθανότητες είναι ανοιχτέ, αλλά πάντα υπάρχει και συζήτηση με τα κράτη-μέλη. Γιατί τελικά η εφαρμογή του νομικού εργαλείου για, τα, για το εμπόριο είναι μια απόφαση την οποία θα τη λάβει το Συμβούλιο, όχι εμεί, όχι ούτε το Κοινοβούλιο, ούτε η Επιτροπή. Είναι απόφαση του Συμβουλίου. Επομένω, σίγουρα δεν μπορούμε να αντιταχθούμε στην άποψη που εκφράζει το Συμβούλιο. Σα παρακαλώ αυτό να το καταλάβετε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ γρήγορα. Μισό λεπτό κύριε Γκάλαχερ. Δέκα δεύτερα, πρέπει να τελειώσουμε. Ο κύριος Γκαλαχέρα έκλεισε το μικρόφωνο του όμως. Οι υπηρεσίε είπαν στο γραφείο μου 10 η ώρα το πρωί ότι δεν πρόκειται να πάρουμε ηλεκτρονικά το έγγραφο. Να πάμε στον Περλεμόντ να το πάρουμε τυπωμένο. Ε, αυτή είναι αλήθεια. Ε, ε, ζητώ συγγνώμη, λυπάμαι. Μπορείτε να λυπάστε όσο θέλετε. Αλλά ε, έτσι έχουν τα πράγματα. Και να κοιτάξετε τις κυρώσεις. Ε, δεν ήταν σωστό ότι θα πάτε στο τέταρτο στάδιο και τώρα ε, τα ρίχνετε στο Συμβούλιο. Κρύβεστε πίσω από τις χώρες μέλη. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Άγνιου, 12. Κυρία Επίτροπε, δεν νομίζω ότι απαντήσατε την ερώτησή μου για τις κυρώσεις κατά των ε, νήσων Φεροέ, αν δεν συμφωνήσουν για τα παράπλευρα αλλιεύματα. Ναι. Ναι, πράγματι, το παρέλειψα. Ελπίζω οι νήσοι Φερός και εμείς να συμφωνήσουμε και το ελπίζω διότι ήμουνα σε επαφή μαζί τους και έχω ήδη πληροφορίες προς αυτή την κατεύθυνση. Αν δεν επέλθει η συμφωνία, η διαδικασία κυρώσεων υπάρχει. Δεν έχουμε αποσύρει τη διαδικασία κυρώσεων, κύριε Άγνιου. Υπάρχει η διαδικασία. Υφίσταται. Ελπίζω να αποσύρουμε μόνο αν επέλθει η συμφωνία με τις Φερόες Νήσους. Είναι σαφές τώρα. Ελπίζω να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Επίσης θα ήθελα να πω ότι εμείς δεν λάβαμε ε, καμία, ε, κανένα έγγραφο από τη Γραμματεία της Επιτροπής μέχρι τις 10.30. Ο κύριος ε, Λεβαντόφσκι κατά την Προεδρία μας είπε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση και ούτε και η Γραμματεία έλαβε κάποιο έγγραφο. Αυτό θα ήθελα να παραμείνει σαφές στο μέλλον να με καλείτε. Έχετε τα δικά μου τηλέφωνα. Εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ. Απλώς θα θέλαμε να πληρούνται όλοι οι όροι όπως πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πίτρο. Ζητώ συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος. Η Επίτροπος φεύγει αλλά η Επιτροπή δεν έχει τελειώσει. Έχουμε και άλλα θέματα γρήγορα. Eh, Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, στα διάφορα υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει ανακοινώσεις του Προέδρου για τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές. Ξέρετε τις αποφάσεις, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Στα διάφορα υπάρχει κάτι άλλο. Όχι. 13. Ανακοινώσεις του Προέδρου για τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές. Όλοι έχετε τις αποφάσεις, ελπίζω να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα προσεχή συνεδρίαση 7 Απριλίου. Μόνο το πρωί. Μόνο το πρωί, όχι πρωί και απόγευμα. Άρα δεν θα συνεδριάσουμε το απόγευμα, μόνο το πρωί της 7ης Απριλίου. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ ο Πρόεδρος και τους ε, διερμηνείς. Γεια σας.